των δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Επίτροπε κύριε Πετώση. Ε, έχουν υποβληθεί τα ψηφίσματα που θα ψηφίσουμε στο τέλος της συζήτησης. Το επόμενο θέμα είναι η Νότιος Κορέα. Η θανατική ποινή κρίνεται παράνομη. Θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στους συντάξαντες. Στάλφος δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά 13 χρόνια χωρί καμία εκτέλεση στην Νότιο Κορέα, είναι πολύ λυπηρό που το Συνταγματικό Δικαστήριο απευθυνθεί υπέρ τη ε, κανονική πηγή. Λένε ότι είναι μία ποινή όπω και οποιαδήποτε άλλη. Είναι κοινό επιχείρημα αυτό και αναφέρεται στην ε, κατάσταση μιας χώρας σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι ε, όταν θεωρείται η θανατική πηγή είναι προληπτικό μέτρο. Κάποιος που θέλει να πράξει μια, ένα έγκλημα που οδηγεί στη θανατική πηγή θα το σκεφτεί δύο φορές. Ναι. Δεν είναι πολύ λογική ιδέα αυτή. Επίσης αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει περιθώριο σφάλματος γιατί μία εκτέλεση είναι αναντίστρεπτη. Έχουμε... Αυτό βασίζεται στον ε, νόμο της εποχής του Ιουσουνιανού, δηλαδή εδώ και 1500 χρόνια. Η θανατική ποινή μπορεί να είναι αντικείμενο σφάλματος και γι' αυτό ε, τα δημοκρατικά όργανα στην Κορέα θεωρούν ότι θα πρέπει να καταργηθεί αυτή η μορφή ποινής με την ένταξη στη Σύμβαση για τα Πολιτικά Δικαιώματα του 1990 και το να είναι τμήμα των περισσότερων ε, συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα ήταν φοβερό για την ε, Νότιο Κορέα να κινηθεί προς τα πίσω. Ευχαριστώ ευχαριστώ κύριε Βέβερ. Ενάμιση λεπτό συνάδελφο Μάτιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα και το Ευρωκοινοβούλιο μα ειδικότερα έχει μεγάλη παράδοση καταπολέμησης και αντίταξης στην ποινή του θανάτου. Και δεν μπορούμε παρά το ίδιο να κρίνουμε και για τη Νότια Κορέα. Παρά το ότι η επιβολή της θανατικής ποινής δεν παραβιάζει το σύνταγμά της. Πρέπει όμως να δούμε τα πράγματα αναλογικά. Την τελευταία φορά που επιβλήθηκε θανατική ποινή επιβλήθηκε με πέντε ψήφους υπέρ και 4 κατά, την προηγούμενη όμως με εφτά ψήφους υπέρ και 4 κατά. Έχει γίνει λοιπόν κάποια πρόοδος και μπορεί κανείς να προβλέψει ότι θα καταργηθεί. Επίσης η Νότια Κορέα είναι de facto χώρα που δεν εφαρμόζει θανατική ποινή από το από εδώ και πολλά χρόνια. Και το 2007 η διεθνή Αμνηστία θεώρησε την Κορέα ως χώρα που πρακτικά έχει καταργήσει τη θανατική ποινή. παρόλα αυτά, όταν βλέπουμε ότι ο αρχηγός του μεγαλύτερου εθνικού κόμματος στην Κορέα Grand National Party θεωρεί ότι πρέπει να επιβάλλεται η θανατική ποινή αυτό σημαίνει ότι πρόκειται τουλάχιστον για οπορτουνισμό. Ελπίζουμε η Νότια Κορέα εκτός από de facto να γίνει και de jure χώρα που δεν εφαρμόζει τη θανατική ποινή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε Μάρτεν. Ο επόμενος για ένα λεπτό συνάδελφος Κάσλερ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι λυπηρό που πολλές χώρες σήμερα στον τον κόσμο εξακολουθούν να χρησιμοποιούν μία απάνθρωπη μέθοδο ποινή σε βαρούς εγκληματίες. Κατά γνώμη μου κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει για την ζωή ενός άλλου ανθρώπου είτε στην αρχή της ζωής του είτε στο τέλος και ούτε όταν πρόκειται για ποινή για κάποιο έγκλημα αυτή η βαρβαρική ποινή της εκτέλεσης δεν έχει θέση στη στο σημερινό κόσμο. Ο Ιωάννης Παύλος ο δεύτερος είχε αναφέρει ότι η ευκαιρία, η δυνατότητα μιας ε, συμφιλίωσης θα πρέπει πάντα να υπάρχει. Αυτό δεν είναι δυνατόν όμως μετά από μια εκτέλεση. Και γι' αυτό καλώ, καλώ τους συναδέλφους στην Νότιο Κορέα να εξάσουν το θέμα αυτό στην Βουλή τους και να αμυνθούμε μαζί μας με τους Ευρωπαίους για ανθρωπιστικούς λόγους για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Και θα ήθελα όλοι οι συνάδελφοι να υποστηρίξουμε αυτή την κοινή πρόταση ψηφίσματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ένα λεπτό, η συνάδελφος Βεζιά. Lors du 4e congrès mondial contre la peine de mort, Κατά το 4ο διεθνέ Συνέδριο κατά τη θανατική ποινή στη Γενέβη ε, εξέφρασαν τη χαρά τους οι σύνεδροι γιατί όλο και περισσότερες χώρες την καταργούν τη θανατική ποινή και η Νότια Κορέα θεωρήθηκε ως στη Νότια Κορέα θεωρήθηκε θετικό ότι επί πολλά χρόνια δεν είχε επιβληθεί θανατική ποινή παρά το ότι νομικά δεν είχε καταργηθεί. Το ότι ξανάρχισε να επιβάλλεται είναι κάτι το οποίο μας λυπεί. Θα έπρεπε η Κομισιόν και το Συμβούλιο να θεωρήσουν τη θανατική ποινή που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ως ουσιώδες κριτήριο για τη σύναψη σχέσεων της Ένωσης με τρίτες χώρες και να ζητήσουν από την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας και τον ίδιο τον πρόεδρο της κυβέρνησης που είχε καταδικαστεί σε θάνατο και ο ίδιος το 81 να ζητήσει την κατάργηση της ποινής αυτής ή τουλάχιστον ένα μορατόριουμ γιατί οι 59 καταδικασμένοι σε θάνατο εξών μερικοί πολιτικοί κρατούμενοι είναι κάτι του σκανδαλώδη. Ευχαριστούμε κυρία Βερζιά. Επόμενος ομιλητής η κυρία Λόχ Μπίλερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η πολιτική για την κατάρριξη τη αντική ποινή είναι ένα επιτυχέ τμήμα τη ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Αυτό φαίνεται σε διαπραγματέ έννοιε, σε διμερεί συζητήσει και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Εθνών. Όσο πάει και περισσότερε χώρε ανά τον κόσμο αποφασίζουν να ε, επιβάλλουν ένα μορατόριο ή να καταργήσουν τελείω την θανατική ποινή. Η Νότιος Κορέα μέχρι τώρα ήταν τμήμα αυτών των χωρών που δεν ε, εφήρμοζαν τη θανατική ποινή. Γι' αυτό αυτή η απόφαση τώρα είναι μια ε, ανησυχητική εξέλιξη και με το ψήφισμά μας θέλουμε να εκφράσουμε την ε, ανησυχία μας αυτή για την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου του Νοτιού Κορέα που δίνει τη δυνατότητα εφαρμογή τη θανατική ποινή εκ νέου. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση στην ε, κυβέρνηση Νοτιού Κορέα να καταβάλει κάθε προσπάθεια καταρχήν για την επιβολή ενό ε, νομικά δεσμευτικού μορατόριου που θα απαγορεύει την, ε, την εκτέλεση. 55 άτομα περιμένουν την εκτέλεσή του, Κατόπιν δε η κυβέρνηση Νοτιού Κορέα θα κάνει καλά να υιοθετήσει ένα νόμο κατά τη θανατική ποινή μέσα στα πλαίσια της ε, κοινωνίας της Νοτιού Κορέας υπάρχει ένα κίνημα που προσπαθεί να συμβάλλει στην υιοθέτηση ενός νομοσχεδίου για την καταδίκηση της ε, θανατικής ποινής. Και αυτούς θέλουμε να τους υποστηρίξουμε εμείς εδώ. Ευχαριστώ, συνάδελφε πιλερ. Εξ πολιτικών ομάδων τώρα, ο κύριος Βαλέζα για ένα λεπτό, εξ ομάδες του. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Νότιας Κορέας είναι εκπληκτική. Η θανατική ποινή θα πρέπει να καταργηθεί και ε, το να παραμένει στο νομικό σύστημα μιας χώρας είναι ένδειξη υποκρισίας. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι δεν μπορεί να, ε, να ανατραπεί. Πρόκειται για μία ε, εκτέλεση και κάποιος στερείται το μοναδικό δικαίωμα που έχει, που είναι η ζωή του. Ταυτόχρονα υπάρχει και ευθύνη για όσους ε, εκτελούν κάποιον ο οποίος είναι αθώος. Για χρόνια στην ε, Νότια Κορέα δεν υπήρχαν εκτελέσεις. Φαντάζομαι, ελπίζουμε ότι η απαρούσα απόφαση δεν θα αλλάξει την κατάσταση και ελπίζουμε ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί η θανατική ποινή. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος ένα ε, ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Νότια Κορέα είναι μια χώρα με την οποία έχουμε πάρα πολλές εμπορικές σχέσεις και είναι μία από τις χώρες που έχουμε διαπραγματευτεί η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου και έχουμε πρόσβαση ο ένας στην αγορά του άλλου. Επομένως, οι εμπορικές μας σχέσεις αποτελούν πρότυπο, είναι πάρα πολύ καλές και αυτή τη στιγμή μας εκπλήσει το γεγονός ότι έχουμε τόσο μεγάλες διαφορές όταν συζητάμε θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τη θανατική ποινή. Η θανατική ποινή θα πρέπει να καταργηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάντα υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής ε, στο διεθνές πεδίο. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να υποστηρίξουμε το κίνημα των πολιτών στην Νότια Κορέα που μάχεται υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής. Ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου να το επιτύχουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποκτήσει νέες εξουσίες ε, στην ε, πολιτική εμπορίου και επομένως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε όλοι οι εταίροι μας να καταργήσουν τη θανατική παινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σνάφας Βασιόπλου έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. αν είχαν εφαρμοστεί οι σημερινέ απόψει για τη θανατική ποινή στη διάρκεια τη δίκη τη ε, Νιρεμβέργη, κανένα από του υπευθύνου ε, για το θάνατο εκατομμυρίων ατόμων δεν θα είχε καταδικαστεί ει θάνατο. Δεν έχω ακούσει ποτέ κανέναν να επικρίνει τι αποφάσει τη δίκη τη Νιρεμβέργη. Η απάντηση σε ένα αδίκημα θα πρέπει να είναι ανάλογη του αδικήματος, του εγκλήματος. Αν μιλάμε για παράδειγμα για γενοκτονία η οποία έγινε στην Ευρώπη, θα πρέπει να υπάρχει και ανάλογη ποινή γι' αυτό. Ευρωπαίοι ακαδημαϊκοί ε, συζητούν και την ε, προληπτική πτυχή της ε, ποινής αυτής. Βέβαια, δεν είναι αυτό το θέμα. Η Ευρώπη έχει καταργήσει τη θανατική ποινή μέσω δημοκρατικών απεφάσεων και θα πρέπει να σεβόμαστε όμω και την άποψη των άλλων επί του θέματο. Εγώ λοιπόν είμαι υπέρ του να γίνει ένα διάλογο με την Νότια Κορέα επί του θέματο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζιώβε. Η κυρία Ρόσπαχ δυστυχώ απουσιάζει. Ολοκληρώσαμε λοιπόν εδώ του ομιλητέ εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων. Ο συνάδελφο Μιγκάλσκι, ένα λεπτό. Oh, sorry. E, panie przewodniczący! Νομίζω ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά της χώρας αυτής για το θέμα αυτό διότι η Νότια Κορέα είναι δημοκρατικό κράτος και το συνταγματικό της δικαστήριο αποφάσισε νόμιμα, νομότυπα δεν υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος αυτή η καταδίκη να εφαρμοστεί, να γενικευτεί. Θα αφορά μόνο σε σημασμένους εγκληματίες και δεχθεί εγκλήματα. Έτσι ώστε η θανατική ποινή να αποτελέσει και αντικίνητρο για την εγκληματικότητα. Αυτό είναι το σημαντικότερο δυνατό αντικίνητρο μάλιστα και μπορεί να σώσει ζωές αθώων. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να παρέμβουν στα εσωτερικά της Νότιας Κορέας για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Άλφα Λουγκάνσκι, περνάμε στη διαδικασία Κασιδιάη. Ο συνάδελφος Σόνικ έχει το λόγο. Dziękuję, panie przewodniczący. Ze smutkiem trzeba przyjąć orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Είναι λυπηρή η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Νότιας Κορέας γιατί αποτελεί επαναχώρηση εφόσον η χώρα δεν έχει εκτελέσει κανέναν για τα τελευταία 13 χρόνια. Αναμένονται βέβαια 57 θανατικές καταδίκες. Πρέπει λοιπόν να καταδικάσουμε την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Η Νότια Κορέα είναι ο κύριος εμπορικός παράγων στην περιοχή εκείνη και πρέπει να αποτελεί παράδειγμα και ηθικά. Η θανατική ποινή δεν είναι αντικίνητρο, δεν οδηγεί σε μείωση της εγκληματικότητας. Τέλεια. Ευχαριστώ συνάδελφε Σανή. Ο Σλαφός έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, η θανατική ποινή είναι θέμα που θα τίθεται όσο υπάρχουν τέρατα μεταξύ των ανθρώπων. Διότι πόσα θα μπορέσει η κοινωνία να τιμωρήσει και να σταματήσει τις τερατώδεις τους δραστηριότητες χωρί τη θανατική ποινή. Φαντάζε, φανταστείτε να συναντήσετε ένα τέτοιο τέρας κατά τη διάρκεια της ζωής σας. Έχουν το δικαίωμα τέτοια τέρατα σε δίκαια δίκη. Τα θύματα είχαν καμία δίκαια δίκη. Το γεγονός ότι οι πολιτικές ελίτ δεν δέχονται τη θανατική ποινή δεν σημαίνει ότι έχει βελτιωθεί η κοινωνία ή ότι έγινε πιο ανθρώπινη ή ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των κτηνοδών τεράτων. Δεν πρέπει να, θυμόμαστε, να φοβόμαστε τη θανατική ποινή. Εγώ σέβομαι τα πρότυπά μας αγαπητοί συνάδελφοι, αλλά να μην θέλουμε να τα επιβάλλουμε και σε χώρες σαν την Νότια Κορέα, εάν πρόκειται για καλύτερη λύση, γιατί όχι. Ε, τελευταία στην Κατσουδιά, η κυρία Σιντλίτσκα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιστήσω ότι προσοχή σα στο γεγονό ότι είναι πάρα πολύ λυπηρή αυτή η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Νότιο Κορέα. Η τελευταία εκτέλεση είχε γίνει το 1997 στη χώρα αυτή. Τώρα όμω βλέπουμε μία απόφαση που ορίζει το ότι η θανατική ποινή δεν είναι αντίθετη με τα δικαιώματα για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή σε αντίθεση με το σύνταγμα της χώρας. Το ανώτατο δικαστήριο είπε ότι η κοινωνία είναι υπέρ της θανατικής ε, ποινής. Λυπούμεθα γι' αυτό. Γιατί η Νότια Κορέα είναι ένας οικονομικός ηγέτης στην περιοχή και θα πρέπει να είναι και ένα παράδειγμα για την πρόσφυση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ συνάδελφε Τσιρέσκα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία Καζιάς και ο επίτροπο έχει το λόγο. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η μάχη κατά της θανατικής ποινής βρίσκεται στην καρδιά της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θεωρούμε ότι η θανατική ποινή είναι μια βάναυση, απάνθρωπη ποινή, που τιμωρεί την εγκληματική συμπεριφορά, ενώ η κατάργησή της ε, βοηθά στην ενίσχυση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Χαιρετήσαμε πολλές θετικές εξελίξεις ε, στη μάχη κατά της θανατικής ποινής. Τον Ιανουάριο φέτος η Μογγολία ανέφερε ότι θα ε, ξεκινήσει ένα μορατόριο κατά της θανατικής ποινής. Το 2009 το Μπουρούντι, το Τόγκο και το Μεξικό ανέφεραν ότι θα καταργήσουν τη θανατική ποινή. Και επίσης ε, υπήρξε ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών που καλούσε τα κράτη-μέλη να θέσουν μορατόριουμ για την ε, κατάργηση της θανατικής ποινής, για τις εκτελέσεις, ε, εν ώψη της κατάργησης της θανατικής ποινής. Το 2008 επαναβεβαιώθηκε αυτό το, αυτή η έκκληση με νέο ψήφισμα. Η απόφαση αυτή βέβαια της Νότιας Κορέας ήταν ε, ε, απογοητευτική ε, από το Συνταγματικό Δικαστήριο στις 15 Φεβρουαρίου. Είχαμε ψηφοφορία 5 προς 4 και αποφασίστηκε ότι αυτό συνάδει με τις διατάξεις του Συντάγματος. Βέβαια ξέρουμε ότι αυτό αφορά στην ερμηνεία του Συνταγματικού Δικαστηρίου στη Κορέα. Δεν έχει να κάνει με την αυτή καθεαυτή εκτέλεση της ανατικής ποινή. Επίσης ξέρουμε τις απόψεις που εξέφρασαν οι τρεις από τους πέντε δικαστές που θεωρούν ότι αυτό συνάδει με το Σύνταγμα. Ο δικαστής Λίκεν Κοκ και ο δικαστής Μιν Χιαν διευκρίνησαν ότι υπάρχει ανάγκη να περιοριστεί η χρήση της θανατικής ποινή και να ε, περιοριστεί και ο αριθμός των αδικημάτων τα οποία έχουν ως ποινή τη θανατική ποινή. Οποιαδήποτε απόφαση για θανατική ποινή θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο δημόσια συζήτησης και απόφασης από τον νομοθέτη. Παρά το γεγονός ότι τα δικαστήρια εξακολουθούν να επιβάλλουν θανατικές ποινές, το, η Νότια Κορέα έχει ένα μορατόριο για τις εκτελέσεις από το 1997 και δεν υπάρχει καμία ένδειξη προς το παρόν ότι η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου θα επηρεάσει το μορατόριο. Είμαστε υπέρ λοιπόν της αποφασιστικότητας της Νότιας Κορέας να διατηρήσει το μορατόριο για τις εκτελέσεις και επειδή ε, το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών έχει πει ότι τα μορατόρια δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως το τέλος αυτό καθεαυτό, θα πρέπει να θεωρούνται η άγουσα προς την ε, τελική κατάργηση. Γι' αυτό λοιπόν παρακινούμε την Εθνική Συνέλευση της Νότιας Κορέας να λάβει βήματα προκειμένου να καταργηθεί οριστικά η θανατική ποινή ε, διότι η Νότια Κορέα ήταν από τις χώρες οι οποίες ε, προσπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Νότιας Κορέας ε, στην προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ, Επίτροπε Πετώσνη. Πέντε ψηφίσματα έχουν υποβληθεί για το θέμα αυτό. Κλείνει η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει τώρα. Αρχίζουμε με την περίπτωση της Λατσάρη. Υπάρχουν ε,